Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε. Συγγνώμη, Μπάρμπαρα. Καλησπέρα σας και πάλι. Έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα στην απογευματινή ημέρη σε διάταξη. Πρώτα θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης, ε, κυρίως τις τροπολογίες, το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Παρβάνοβα, που θα δώσουμε στην Επιτροπή Γυναικών και στην Νομική Επιτροπή με θέμα την πρόταση οδηγία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Η κυρία Παρβάνοβα είναι η συγγήτρια, ε, για το ε, ΕΛΚ. Εγώ είμαι σκιώδης ε, και μάλιστα μόνο ως άνδρας σκιώδης ηγητής από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικού και ε, έχουμε γυναίκα επίσης εκπρόσωπο από τους σοσιαλιστές. Χωρίς άλλη καθυστέρηση να δώσω το λόγο στην κυρία Παραβάνοβα για να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες. Και αν δεν κάνω λάθος, ε, έχουν συνταχθεί κάποιες συμβαστικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους και οδησηγητές και όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες. Να τους ευχαριστήσω θερμά για το έργο τους και κυρίως σε τους και οδησηγητές γιατί ε, συνέβαλαν στην εξισορρόπηση της γνωμοδότησης και στην καταπράση των πνευμάτων ε, στην Επιτροπή για ένα τόσο επίμαχο θέμα. Γενικώ η οδηγία δεν είναι τόσο επικίνδυνη και τοξική αν καταφέρουμε και βρούμε μια συνετή προσέγγιση και ισορροπημένη και θα πρέπει να περιοριστούμε στι αρμοδιότητε τη επιτροπή μα. και να αναζητήσουμε μια ισορροπημένη λύση που θα εξυπηρετεί όλου και χωρί να δημιουργεί αντιφάσει, θα ανταπεξέρχεται στι προσδοκίε μα. 66 τροπολογίε κατατέθηκαν συνολικά, από τι οποίε συντάξαμε 6 συμβαστικέ τροπολογίες. Η πρώτη συμβαστική τροπολογία είναι εύκολη, αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αντίκτυπο των ε, επιλογών των γυναικών ε, και την επιρροή τους ε, στην, στις δαπάνες των καταναλωτών. αναφέρεται σε μια δική μου τροπολογία και μια τροπολογία της κυρίας Λεγκρίπ. Είπαμε να μιλήσουμε για γενική περιγραφή του συνόλου των καταναλωτικών δαπανών που ελέγχονται από τις γυναίκες. Αυτή πάντως ε, είναι μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια απλή παραπομπή σε αυτή δεν προβληματίζει γιατί τόσο άλλως πρόκειται για επίσημη μελέτη. Η δεύτερη συμβαστική τροπολογία αναφέρεται στην ευθύνε μας και στη μέρημνά μας ε, για τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείε να λαμβάνουν υπόψη, φυσικά να λαμβάνονται αυτές οι διαδέξεις υπόψη και από τα θεσμικά όργανα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί και εκεί διαπιστώνονται ανισορροπίες ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των φύλων. Προτάθηκε να μην κατονομαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να μην αναφερθεί ρητά, παρά την αντίθετη τροπολογία κάποιων συναδέλφων. Εγώ συμφωνώ ότι αν αρχίσουμε να κατανομάζουμε τα θεσμικά όργανα δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε ορισμένα από αυτά, θα πρέπει να τα αναφέρουμε όλα ονομαστικά. Υπάρχει αρκετά, αρκετή διάσταση απόψεων στο Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκε ότι ε, η πρόταση για το, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το της ΕΚΤ ε, δεν γίνεται σεβαστή από το Συμβούλιο. Πάντως, αν αναφερθούμε σε ε, κοινοτικούς ενωσιακούς οργανισμούς, θα πρέπει, αν είναι να κατονομάσουμε την Κεντρική Τράπεζα, να κατονομάσουμε και άλλες, αλλιώς η ψηφοφορία για να μην υπάρχει πρόβλημα. Συμβαστική τροπολογία 3. Ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να διαδίδουν τις ευέλικτε πρακτικές. Στερεότυπη διατύπωση. Ενθάρρυνση των κρατών μελών για ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Δεν είναι πρόβλημα γιατί τους άλλους είναι προαιρετική αυτή η δυνατότητα. Συμβαστική τροπολογία 4. Τροπολογίες Χάν, Χάρμπορ και Μάντερς. Αφορά τη χειρία κάποιων θέσεων και της, ε, την πρόταση για υποβολή υποψηφιωτήτων. Αφορά ε, και την τροπολογία 6 που μιλάει για τα κριτήρια αυτής της κένος και των διαγωνισμών μετά από αυτές. Και τέλος, συμβαστική τροπολογία 5 που θα χαροποιήσει ακόμη και τους πιο σκεπτικιστές συναδέλφους για το θέμα αυτό, γιατί αναφέρουμε στην τροπολογία αυτή ότι θα πρέπει να σεβόμαστε το οικονομικό και νομικό πλαίσιο των κρατών μελών αυτή η συμβαστική τροπολογία 5 στηρίζεται σε αντίστοιχε τροπολογίε των Harbor και Le Αυτά ω προ τι συμβαστικέ τροπολογίε. Ελπίζω να συμφωνείτε με την ισορροπημένη επιλογή που έκανε αυτή η γνωμοδότηση, να την υπερψηφίσετε και να μην ξεφύγουμε από τι συμβαστικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ, κυρία Παρβάνουβα. Σας ευχαριστώ που συντάξετε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Πολύ καλή δουλειά. Έχουμε τους κοιόδης εισηγητές ε, τώρα και εν συνεχεία θα ακούσουμε τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Ε, η κυρία Λεγκρότη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγητριά μας για τη δουλειά που έκανε της γνωμοδότησης. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ισορροπία στην εκπροσώπηση των γυναικών ε, σε θέσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις και κυρίως οικονομικές αποφάσεις. Να υπενθυμίσω σύντομα ότι στις προηγούμενες παρεμβάσεις ε, του ΕΛΚ είχαμε υποστηρίξει συνολικά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μέσω της πρότασης οδηγίας επικοδομητικό πνεύμα, δείχνει η Επιτροπή εκεί. Είναι πολύ και φιλόδοξη, αλλά και ευέλικτη, ισορροπημένη. Και χαίρομαι που αυτό το πνεύμα ευελιξίας, ρεαλισμού, αλλά και θέλησης, απεικονίζεται στο κείμενο της εισηγήτριας, στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης με το οποίο ταυτιζόμαστε, με τις απόψεις το ταυτιζόμαστε. Ε, εξ ονόματος ομάδας μου θα υποβάλω α, κάποιες τροπολογίες, ούτως ώστε οι αρμοδιότητες των γυναικών να κρίνονται και να αξιολογούνται όπως ακριβώς των ανδρών. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσουμε ούτως ώστε η διαδικασία επιλογής να είναι δίκαιη, διαφανής, να υπάρχει ισοτιμία γιατί νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, εκεί έγκυται η έλλειψη ισότητας στις κοινωνίες μας. Το σχέδιο, της συμβαστικές τροπολογίες μπορούμε να τις υποστηρίξουμε εκτός ε, από την συμβαστική τροπολογία 2. Αν δούμε λίγο την ε, διατύπωση της, ε, μας δημιουργεί κάποια προβλήματα. Ζητώ συγγνώμη που παρά τις ε, διαπραγματεύσεις που κάναμε δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε όλες οι ομάδες. Εμείς είπαμε ότι ζητάμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Αν ικανοποιηθούμε εκεί, με τη χωριστή ψηφοφορία, με ψηφοφορία κατά τμήματα δηλαδή, θα μπορούσαμε τελικά να συμφωνήσουμε με το κείμενο όπως θα προσαρμοστεί για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή της παρούσα οδηγίας και η τεχνική κατονόμαση ενό θεσμικού οργάνου δεν νομίζω ότι είναι και πολύ επιτυχημένη. Εντάξει, να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. να μπορούν και αυτά να μπορούν να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη το ρόλο των γυναικών και τις γυναίκες στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, να μην κατανομάσουμε ένα συγκεκριμένο θεσμικό όργανο, δεν είναι σωστό. Για τις άλλες τροπολογίες των άλλων συναδέλφων. Είναι σαφής η θέση μας. Η γραμμή μας είναι ότι θέλουμε να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές και στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Απορρίπτουμε κάθε τροπολογία που αποδυναμώνει ή που ενισχύει υπερβολικά τις διατάξεις της ε, πρότασης της οδηγίας ή που τις αποδυναμώνει λοιπόν ή που θέλει να διευρύνει τις αρμοδιότητες ή το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Η ομάδα του ΕΛΚ δεν θα υποστηρίξει επίσης τις τροπολογίες 6 και 56 που σκοπό έχουν να καταργήσουν τον, ε, την εξαίρεση των ε, επιχειρήσεων που έχουν λιγότερο από το 10% του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Δεν θα υποστηρίξουμε αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σκεφτούμε λιγάκι τα όσα διαμείβονται σε αυτή την Επιτροπή. Κανονικά η Επιτροπή μας είναι γεμάτη από άντρες με κουστούμια, ε, αλλά σήμερα ε, το πράγμα έχει αντιστραφεί. Έχουμε δύο θαραλέους έτσι, άντρες με κουστούμια και τις κομψές κυρίες. Αν δούμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και την ισότητα των φύλων και πώς εκφράζεται, σκέφτομαι ότι οι άνδρες στην Επιτροπή μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Με απογοητεύει αυτό. Με απογοητεύει που δεν είναι περισσότεροι άνδρες. Πρέπει να το πω αυτό. Να το βγάλω από πάνω μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία. Έκανε θαυμάσια δουλειά. Έκανε πραγματική προσπάθεια ούτως ώστε να λάβει υπόψη όλους μας ε, στις συμβαστικές τροπολογίες και με ικανοποιεί αυτό. Τώρα, κάποια θέματα που θέσαμε εμείς οι σοσιαλδημοκράτες και που για μας είναι κόκκινες γραμμές. Καταρχάς, αυτή η ανοιχτή διαδικασία αναζήτησης νέων μελών ενός Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να μπορούν και οι γυναίκες να κάνουν κάτι όταν αισθάνονται ότι υπάρχουν διακρίσεις εναντίον τους. Είναι πολύ σημαντικές οι κυρώσεις και οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι σκληρές. Γιατί αλλιώ δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Θα είναι απλώ ε, χειρονομία, χειρονομία κενή περιεχομένου αν δεν έχουμε και κυρώσει. Υπάρχει και ένα άλλο λεπτό θέμα που έχει ζητηθεί αρκετά. Θέλουμε η Κομισιόν να εξετάσει τη δυνατότητα των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Και αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία, από αυτό το νομοθέτημα. Αυτό πιστεύουν οι σοσιαλδημοκράτε. Και ελπίζουμε να γίνει μια καλή ψηφοφορία αύριο. Η κυρία Ρούλε, Θέλει και αυτή να πάρει το λόγο. Ρούλερ. Äh, Πατάω το λάθος κουμπί. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστώ τον, ε, την εισηγητρία για την πρόταση και τις συμβαστικές τροπολογίες. Την υποστηρίζουμε πλήρως. Προφανώς δεν και δυστυχώς δεν σας υποστηρίζουν όλα τα μέλη της ομάδας σας. Λυπούμε γι' αυτό. Αλλά, εν πάση θα δούμε. Και ο κύριος Ροσφόρ είναι εδώ. Ο κύριος Μάντερς βλέπουμε πόσες τροπολογίες έχει κάνει και άλλοι συναδελφοί σας αποδυναμώνοντας το κείμενο. Ίσως μπορούμε να το συνασύστησουμε κάποια άλλη στιγμή. Πάντως σας υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Χέιντι, είμαι παρόν όχι μόνο ως Πρόεδρος, αλλά και γιατί θέλω πράγματι πολλές γυναίκες να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο θέσεις ηγετικές. Υπάρχει αυτό που λέμε σε πολλέ εταιρείε τουλάχιστον ε, γυάλινη οροφή πάνω από την οποία δεν μπορούν να αρθούν. Εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή μπορεί σε ένα πολύ μικρό τομέα στις ε, ενταγμένες ε, στο χρηματιστήριο εταιρείε να κοιτάξει, να υποστηρίξει αυτή την παρουσία των γυναικών. και η κυρία Παρβάνοβα έχει κάνει πολύ καλές και χρήσιμες αλλαγές. Μπορούμε να δεχθούμε τις συμβαστικές της τροπολογίες και γενικότερα την προσέγγιση της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιτρέψει χώρες που είχαν διαφορετικές μεθόδους, όχι μόνο νομικές για την πρόθεση των κινητών γυναικών σε αυτές τις θέσεις, να συνεχίσουν να το πράττουν. Και βεβαίως καλά κάνει σε έναν βαθμό. Ε, δεν χρειάζεται πάντοτε να έχουμε νομοθετικά μέτρα. Όταν αυτά φέρουν αποτέλεσμα, όταν τα μη νομοθετικά φέρουν αποτέλεσμα, βέβαια, γιατί στην Νορβηγία είδαμε ότι φέρουν αποτέλεσμα, αλλά εκεί ίσω ήταν λιγότερε δυσκολίε. Πάντω βλέπουμε ότι όταν έχουμε γυναίκε σε διοικητικά συμβούλια, αλλάζει και ολόκληρη η νοοτροπία και η συμπεριφορά μια επιχείρηση και ο τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσει ε, τα διοικητικά συμβούλια. Και ιδιαίτερα το βλέπουμε αυτό σε μεγάλε εταιρείε. Γιατί πρόκειται μάλλον για θέμα και νοοτροπία. Δεν είναι μια απλή αλλαγή, δηλαδή είναι πολύ πιο βαθιά η αλλαγή του να μπουν και γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Λυπούμε που δεν υπάρχουν πιο πολλοί συνάδελφοι, όπως είπε και η κυρία Χέιντι, να το συζητήσουμε. Πάντως, στο δημόσιο τομέα και χωρίς να έχω δει στοιχεία αναχώρα, μάλλον έχουν καλύτερες επιδόσεις στο δημόσιο σε ηγετικέ θέσει. Οι γυναίκες. Και υπάρχουν ε, θεσμικά ζητήματα. Εργοδότες ε, οι οποίοι ευνοούν περισσότερο τις γυναίκες, αξιολογούν ε, πιο καλά τις επιδόσεις τους και το καθεξές. Αν λοιπόν μου ζητηθεί να βελτιώσω την κατάσταση, θα πρέπει να κάνω συγκριτικές ε, μελέτες και για τα θεσμικά όργανα βεβαίως και για τις μεγάλες θετικές επιχειρήσεις και ίσως να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων ε, στο δημόσιο του Ηνωμένου Βασιλείου το τρέχει μια γυναίκα, την οποία γνωρίζω πολύ καλά. Ήταν άλλωστε επικεφαλής και στις τοπικές αρχές της ε, δικής μου περιφέρειας. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει αναγνώριση και ανέλυξη γυναικών στο δημόσιο κυρίως. Χρήσιμα λοιπόν το είπε η κυρία Παρβάνοβα, την ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε και προς το έργο της Επιτροπής των Γυναικών, διότι σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την επικοινωνία μαζί τους. Και ξέρω ότι κάνανε ένα σχόλιο ως προς το ότι οι γυναίκες λαμβάνουν απόφαση ως καταναλωτές, έχουν κύριο ρόλο να λαμβάνουν αποφάσεις ως καταναλωτές και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Και ίσως αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει περαιτέρω. Αυτή ήταν η δική μου η συμβολή ως και όδου ηγητού εκ μέρους της ομάδας μου. Και επανέρχομαι στο ρόλο μου ως Προέδρου για να ακούσουμε την κυρία Αμπέλα, την οποία και πάλι καλωσορίζω. Δεύτερη παρέμβαση στην Επιτροπή μας. Σα δίνω το λόγο. Και η κυρία Βάιλερ νομίζω. Η κυρία Μπέλα και η κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η έκθεση Παρβάνοβα έρχεται την καταλληλότερη δυνατή στιγμή. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη δημοκρατία, για τα δικαιώματα, για την ισότιμη εκπροσώπηση της γυναίκας στην πολιτική και οικονομική ζωή που αποτελεί ένα ζήτημα και ένα ζητούμενο για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αναγκαίο κακό θα έλεγα η συζήτηση της έκθεσης. Και το να έχουμε μια πιο ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών σε υψηλότερα επίπεδα έχει σημασία όχι μόνο για την καλύτερη και πιο δίκαιη εκπροσώπησή τους στην κοινωνία, αλλά και γιατί οδηγεί σε καλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα, πιο λογική επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως δείχνουν και μελέτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μελέτησε ακριβώς, μελέτησαν ακριβώς την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις, που παρουσιάζουν αποτελέσματα και περιβάλλον πιο ε, θετικό, πιο καλές επιδόσεις και καλύτερο κλίμα εργασιακό στην επιχείρηση. Οι γυναίκε και οι άντρε που να συμπληρώσω έχουν διαφορετικές εμπειρίες από την ε, διαφορετική κοινωνική αλλά και βιολογική δομή τη ζωή των ε, δύο φίλων και έτσι μπορούμε να έχουμε μια πληρέστερη εκπροσώπηση. Μια καλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των φίλων και στην λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων θα μπορούσε να εισαγάγει τη μικροοικονομική προοπτική μέσα στις επιδόσεις των ε, μεγάλων επιχειρήσεων και όχι μόνο μακροοικονομική, ε, που σημαίνει βέβαια και βιώσιμη ανάπτυξη και ρυθμός ανεκτούς. Και για να μιλήσω για τη Μάλτα, την πατρίδα μου, έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό γυναικών με υψηλή μόρφωση και κατάρτιση. 60% τα πτυχία τον, ε, τα πτυχία κάθε χρόνο τα παίρνουν οι γυναίκες και έτσι δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να βρεθεί μια γυναίκα με σωστή κατάρτιση και δεξιότητες ώστε να αναλάβει καθήκοντα μαζί με τους άνδρες ομολόγους της και συναδέλφους της. Αλλά πάλι πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι διαφορετική η κοινωνική ε, αντιμετώπιση και ανατροφή ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν παγιωμένοι και δρεωμένοι ρόλοι για τα φύλλα οι άντρες μεγαλώνουν μαθαίνοντας να εκπληρώνουν τον ρόλο του ανδρός ή δε γυναίκες της γυναικός. Και πολλές φορές αυτό που συμβαίνει είναι ότι υλοποιούμε αυτό το οποίο έχουμε μάθει ε, μεγαλώνοντας. Το ρόλο δηλαδή που μας έχουν διδάξει. Πρέπει λοιπόν η θέση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και τις ηγετικέ θέσεις για να εξασφαλιστεί να λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες, τις θεωρίες, την κόσμοθεωρία, την πραγματικότητα των γυναικών. Δηλαδή οικονομική, δημοσιονομική, πολιτική, ε, περιβαλλοντική και γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω την έκθεση Παρβάνοδα και τις τροπολογίες της. Thank Σας ευχαριστώ. Κυρία σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μια πολύ μικρή ε, συμπλήρωση μόνο και χαίρομαι ιδιαίτερος, πρέπει να πω, διότι βλέπω ότι όλες οι ομάδες στην Επιτροπή μας συμμερίζονται τη βασική στοχοθέτηση και εσείς ακόμα Μάλκομ που θέλετε να την ξεπεράσετε, να πάτε πιο πέρα ακόμα από αυτή τη στοχοθέτηση. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που το βλέπω. Ε, δεν ξέρω γιατί μα ζητήσε η Επιτροπή Γυναικών τη γνωμοδότηση αυτή, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να την τυπώσουμε. Αποδεικνύεται ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία της Επιτροπής μας ως ε, αρμόδιας για νομοθετήματα Επιτροπής και έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή παρουσία και στην τελική συζήτηση στην Ολομέλεια και τελική ψηφοφορία. Οι γυναίκε δεν θα πω πάντα ότι είναι ο καλύ, οι καλύτεροι, ότι είναι καλύτερες από τους άντρες δηλαδή, αλλά όταν βλέπουμε γυναίκες σε τράπεζες, ε, στο στη βιομηχανία, σε μεγάλε επιχειρήσεις, πώς έχουν χειριστεί υποθέσει και καταστάσεις πολύ διαφορετικά από ότι άντρε, Ίσως να μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αν είχαμε πιο πολλές γυναίκες στους χώρους αυτούς δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την φοβερή και τρομερή κρίση που αντιμετωπίζουμε. Αυτό το έχουν πει πολλοί οικονομολόγοι. Και κάτι ακόμη για το δημόσιο τομέα. Με κατάπληξη βλέπω ότι στις ανώτατε θέσει στον δημόσιο τομέα πάλι δεν είναι πολλέ οι γυναίκε. Δηλαδή δεν είναι πολλέ οι γυναίκε πρωθυπουργοί κρατηδίων, στι ομοσπονδιακέ δομέ ή ε, δήμαρχοι. Από την άλλη όμως, αμέσως κάτω από το επίπεδο αυτό ε, και πάντως με ισότιμο αμοιβή, βλέπουμε πολλές γυναίκες και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία βλέπουμε τουλάχιστον ε, πως έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα της ισότιμης αμοιβή για θέσεις ευθύνη μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μίλης μονούμε επίσης ότι η κυρία Ρέντινγκ, η Επίτροπος, ε, χρειάστηκε πολλές φορές να προβάλλει πρωτοβουλίες και να επιμείνει για την ίδια πρωτοβουλία πολλές φορές μέχρι ότου οι άνδρες ε, συνάδελφοί της, αλλά ίσως και γυναίκες επίτροποι θέλησαν ε, να δουν με καλό μάτι τις προτάσεις της. Ίσως λοιπόν ήταν καλό να έχουμε μια πιο ανοιχτή θεώρηση της προτάσεις των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Έχουμε πρόσωπο της Επιτροπής εδώ. Θα θέλατε το λόγο. Συγγνώμη, έχασα το χαρτί με το όνομά σας. Κύριος Γκόγκλε. Θα είχατε την καλοσύνη να μας πείτε τη γνώμη σας από τη μέχρι τώρα συζήτηση ή αν έχετε άλλα σχόλια ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στο τέλος θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Παραβάνοβα για τα καταληκτικά σχόλια. Αύριο ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Μιχαήλ Γκόντεκ. Είμαι νομομαθής ε, στην ε, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής, αλλά κυρίως την εισηγήτρια για την πολύ ισορροπημένη της έκθεση. Και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που δείξετε στη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο ότι διαφυλάξετε το πνεύμα της οδηγίας, που είναι και φιλόδοξη ως προς τους στόχους της, αλλά και ευέλικτη και ισορροπημένη ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Παρβάνοβα, θα θέλετε να ολοκληρώσουμε με κάποια σχόλια. Ναι, να ευχαριστήσω τους συγγητές και όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση και σχολίασαν τις συμβαστικές τροπολογίες και τις υπόλοιπες τροπολογίες. Θα ήθελα να καθησυχάσω το έλκο ότι στη συμβαστική τροπολογία 2 θα έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα και όσοι είναι κατά το να κατανομάζουμε ρητά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να την εκθέτουμε μπορεί να το, να το ψηφίσει. Μερικές φορές όμως εγώ είμαι υπέρα αυτής της, της προσέγγισης, να κατονομάζουμε δηλαδή είτε κάποιους, παρόλο που έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα στην ε, Ολομέλεια. Σίγουρα δεν θέλω να επιτείνω την τάση, είναι αρκετά επιμαχό το θέμα. Ψηφοφορία κατά τμήματα λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε 6 και 56 για το ποσοστό και τον αποκλεισμό τη ε, εκπροσώπηση των γυναικών ή του στόχου τη οδηγία ε, ε, σε επιχειρήσεις που λιγότερο από 10% των εργαζομένων ε, είναι του άλλου φύλου. Πάντως είχα επιφέσει με επιχειρηματίες και είπαν ότι δεν έχουν πρόβλημα με τη διαδικασία αυτή. Άλλωστε οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι σχετικές ε, αποφάσεις δεν δημιουργούν αντίφαση με τα καθήκοντα των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά τις μη στο χρηματιστήριο εταιρείε, σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα ισχύσει και για εκείνε τις μη στο χρηματιστήριο εταιρείε. Πάντω, συμφωνώ με την κυρία Χέντ ότι στο μέλλον ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία ε, στην ανάλυση μας για το θέμα αυτό, γιατί δεν ξέρουμε και πολλά, σε ό,τι αφορά τα πειθαρχικά μέτρα. Συμφωνώ και εγώ ότι θα προτιμούσα πιο φιλόδοξες προτάσεις, αλλά δεν νομίζω ότι πιο φιλόδοξες προτάσεις θα είχαν μεγαλύτερη υποστήριξη. Προτιμούμε να δώσουμε ενάυσματα στα κρατημέλη και να μην τα αποθαρρύνουμε. Προτιμούμε λοιπόν πρώτα μέτρα με ενάυσματα παρά μέτρα με φόβητρα και κατα, κατασταλτικά για τα κρατημέλη. Για τον κύριο Μάντες που είναι ο συγγετής μας είπαμε ότι θα συνεννοηθούμε. Μου είπε πάντως ότι συμφωνεί με την προσέγγισή μου και θα την υποστηρίξει αύριο στην ψηφοφορία. Καλό σημάδι αυτό δηλαδή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάλυση και τη σύγκριση των εταιριών, συμφωνώ ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια ανάλυση, σίγουρα θα αποφεύγαμε πρακτικές τύπου Lehman Brothers ή κάποιων άλλων εταιρεών. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξη και ευελπιστώ ότι αύριο η ψηφοφορία θα είναι αίσια και θα καταλήξει σε έγκριση της γνωμοδότησης. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν στη ψηφοφορία. Και να περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι εξίσου σημαντικό. Επίσης πρόκειται για νομοθετική έκθεση, στην οποία είμαστε και η καθήλια αρμόδια επιτροπή, με θέμα την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. Η συγκήτρια είναι η κυρία Βάιλερ και ο κύριος Βαντερκάμπ είναι σκιώδης για το ΕΛΚ. Ο κύριος Μάντερς απουσιάζει. Ο κύριος Ροσφόρ θα τον αντικαταστήσει για το ραδιοεξοπλισμό ή δεν είστε αρμόδιος. Ή μήπως ο κύριος Μάντερς θα ε, διακτηνιστεί από κάπου στη συνεδρίαση. Κυρία Ρούλε, ο συνήθως είναι σκιώδης για πολλά και διάφορα θέματα και για το συγκεκριμένο. Και να καλωσορίσω και πάλι τον κύριο Ζηράο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον έχουμε δει σε θέματα εποπτείας αγοράς, νέο νομοθετικό πλαίσιο. Θα μας δώσει τη γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. κυρία Βάιλερ ε, προχώρησε με ταχύ ρυθμού σε ό,τι αφορά την εκπόνηση του σχέδιου της έκθεσης. Έχουμε ήδη τι τροπολογίε. Θα ακούσουμε πρώτα την εισηγήτρια, μετά του και του εισηγητές, κατόπιν την Επιτροπή και θα δούμε τη μέλη ενέστη για τη συνέχεια. Κυρία Βάιλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Λεγκρίπ, σας παρακαλώ με ενοχλείτε. θα είμαι σύντομη. Διότι έχουμε ήδη συναντηθεί με τους ε, σκιώδης μια φορά και έχουμε προσδιορίσει ως εκ τούτου την κύρια γραμμή των προτάσεών μας και έχουμε δει και σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και την έγκριση της εκθέσεως Ρόιτοβα η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι στο, στη δική μας γραμμή Εγώ θεωρώ κατά βάση ότι είναι καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στον εξυγχρονισμό ή την προσαρμογή για τα μηχανήματα, ραδιοεξοπλισμό και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσει να αυξάνεται η χρήση τους. Χρειάζεται βέβαια να αφήσουμε περιθώριο και να δώσουμε όθηση στη δημιουργία νέων και καινοτόμων προϊόντων και βέβαια θέσεων εργασίας, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος των ε, παρεμβολών μεταξύ των διαφορετικών προϊόντων, καθώς πρόκειται για ένα τομέα παρουσιάζει όρια λόγω της τεχνολογίας, τεχνολογικά όρια. Έτσι λοιπόν πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, πρέπει να προτείνουμε λύσεις και απλούστευσης ε, της νομοθεσίας και της υλοποίησής της για τον κατασκευαστή. Έχοντας συνομιλήσει με μια σειρά από ομάδες ενδιαφέροντος, συμφερόντων, του τα λόμπι όπως τα λέμε, και χωρίς να εκπροσωπώ κανενός ε, την ε, προτίμηση. Ε, προτιμώ τι θέσει επιτροπή πρέπει να σας πω, οι οποίες μου φαίνονται εν γέννη πιο σωστέ, αλλά σε ορισμένα σημεία θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε και δει εκεί όπου μιλούμε για το σύστημα της καταχώρησης, γιατί δεν έχουμε συμφωνήσει, ίσως και δεν έχουμε πει ακόμα τελευταία μας λέξη στην υπόθεση αυτή. Κατά βάση, θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι και για τον καταναλωτή είναι σκόπιμο να έχουμε μία απλούστευση. Ίσως και στη συζήτηση με τον Επίτροπο Ταγιάννη θα θυμάστε πως ε, είχαμε σημειώσει ότι θα ήταν πολύ καλύτερο για τον καταναλωτή να έχουμε ένα σύστημα με φορτιστές για το κινητό, τον, ε, το λάπτοπ και τα λοιπά μηχανήματα της καθημερινής ζωής μεταξύ τους συμβατούς και ε, που θα μπορούσε να αλλάξει κανείς εύκολα. Ε, είπε η Επιτροπή ότι θα συνομιλήσει με τους ε, παραγωγούς κατασκευαστές. Είναι κάτι το οποίο ήδη έχει προβληματίσει και τους κατασκευαστές, θα πρέπει να το επαληθεύσουμε να μας πει η Επιτροπή εάν όντως είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν οι κατασκευαστές και αν, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, δεν είναι διατεθειμένοι, τότε θα πρέπει να επιβληθεί υποχρεωτική η, ε, η διάταξη αυτή. Ε, δεν το κάναμε ακόμα γιατί ο Επίτροπος μας βεβαιώσει ότι θα βρει μια λύση σε εθελοντική βάση. Διαφορετικό όμως θα πρέπει να επιβληθεί. Ε, και κάτι άλλο, μεγάλο θέμα, παλιό θέμα, δεν καινούριο, στο Κοινοβούλιο, η κατεξουσιοδότηση νομοθετικές πράξεις και εκεί και με την ευκαιρία των άλλων εκθέσεων θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε μια καλή λύση στο Κοινοβούλιο με απλούς κανόνες ε, για τα τεχνικά ζητήματα ασφαλώς δεν θα υπάρχει πρόβλημα αλλά όπου υπάρχει ζήτημα πολιτικής αποφάσεως δεν είμαστε διατεθειμένοι να αναθέσουμε την απόφαση σε τεχνοκράτες και μόνο. Δεσμευτικά συστήματα καταχώρησης. Είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πώς θα το ρυθμίσουμε. Εγώ προσωπικώς και εκ μέρους ομάδος μου θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ δεσμευτική και δεν προσφέρει προσθέμενη αξία, περιπλέκει μάλλον τα πράγματα. Θα προτιμούσα να ακούσω και άλλες γνώμες. Προς το παρόν. Αυτό που βλέπω μόνο να επιδεινώνει την κατάσταση και να περιπλέκεται. Η επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σοβαρή παρουσία στην αγορά και, πλη, και πολλούν τα προϊόντα τους, τόσο άλλο στηρούν αυτές τις προδιαγραφές της ε, καταχώρησης και κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει προσφέρει τίποτα περισσότερο. Στο θέμα της μετάφρασης των δηλώσεων ε, συμμόρφωσης, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε χωρίς προβλήματα. Δεν χρειάζονται 22-23 γλώσσες για μετάφραση. Απλώς χρειάζεται στο εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για το καταναλωτή να υπάρχει μια σαφής γλώσσα, να μην είναι δηλαδή πολύ περίπλοκα τεχνικά στοιχεία, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να βρει ε, χρήσιμη, χρήσιμες πληροφορίες χωρίς περιττή και τεχνοκρατική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που πρέπει να κάνουν τη μετάφραση. Αυτά λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε καλή συνεργασία, ίσως και οι συνάδελφοι σκιώδεις συγητές μπορούν να προσφέρουν κάτι επιπλέον. Μια-δύο τροπολογίες εγώ προσωπικώς μόνο. Πάντως ε, θεωρώ ότι είναι μια καλή προσέγγιση για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση της αγοράς ε, ραδιοεξοπλισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ πολύ θερμά την κυρία Βάιλερ για τον τρόπο, τον καθαρά γερμανικό με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτό το θέμα, που σημαίνει αποτελεσματικό δηλαδή. Από την άλλη, απογοητεύτηκα λιγάκι, γιατί πώς θα κάνουμε πολιτική συζήτηση και θα δώσουμε πολιτική μάχη όταν υπάρχουν τόσο συγκλίνουσε απόψεις. Αλλά τι να σας πω κι εγώ, τεχνικό είναι το θέμα, ίσως είναι και λογικό αυτό. Η έκθεση της κυρίας Βάιλερ Ε, είναι μια έκθεση που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί ως ΕΛΚ έχουμε πολύ στενή σχέση με τον κλάδο. Και η έκθεση Βάιλερ ε, έτυχε θέρμης υποδοχής από τον κλάδο. Φυσικά θα καταθέσω κάποιε τροπολογίε. Η 5η Ιουνίου δεν είναι μια ημερομηνία πολύ μακρινή. Δεν πρόκειται βέβαια να αναδιατυπώσουμε άρδιν την έκθεση με τις, μέσω των τροπολογιών. Το μόνο που θέλω να ρωτήσω είναι τι γίνεται με το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Μιλάμε για κλάδους που λειτουργούν όπως, λίγο, όπως και ο κλάδος των μικροκυμάτων. Ε, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η οδηγία αφορά τους παραλήπτες, τους χρήστες. Δεν αφορά καθόλου τα εξαρτήματα των, του εξοπλισμού αυτού ε, τους έχουμε αφήσει λίγο έξω. Αυτό είναι το σχόλιο που θέλω να κάνω στο πάνω και σε ευχαριστώ κατά τα άλλα. Κυρία Ρούλερ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την κυρία Βάιλερ με τη σειρά μου. Ε, υποστηρίζουμε την έκθεσή τη. Δεν νομίζω να καταθέσουμε πολλές τροπολογίε αν καταθέσουμε καμία. Παντώ υποστηρίζω τη δική σα τροπολογία την 27 για την υποχρεωτική καταχώρηση και εγώ θεωρώ ότι είναι περιττή αυτή ε, και συμφωνώ με την διεύρυνση ως προς το πεδίο εφαρμογής ώστε να έχουμε και τα μηχανήματα λήψης τους δέκτες. Αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει προβλημά και ότι χρειάζονται πολλές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή και ταχύ επεξεργασία του θέματος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Ρούλε. Και εγώ θα είμαι σύντομο γιατί η κυρία Βάιλερ έκανε τις κρίσιμες στρατηγικές αλλαγές και νομίζω ότι πρόλαβε αυτά που θέλαμε να πούμε οι υπόλοιποι και να πετύχουμε οι υπόλοιποι. Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν πρέπει να καταχωρούμε τα, τα προϊόντα. Και επίσης πρέπει να κρατήσουμε ουσιαστικά την ε, σημερινή δομή. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο υπάρχουν ε, και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες που θα παίξουν ρόλο ε, και από τις συζητήσεις του τριμερούς διαλόγου που είχαμε την κυρία Ράιτοβα Ρόιτοβα, ε, μπορούμε να δούμε ποια είναι τα βασικά σημεία. Θα μπορούσαμε οι σκιώδε να τα ξαναδούμε όλα αυτά τα θέματα, ούτω ώστε να σταθούμε στα βασικά. Υπάρχουν τα θέματα της επισήμανσης, η ηλεκτρονική επισήμανση που υπάρχει τώρα στα smartphones ε, και μας δίνει όλες τις πληροφορίες. Δηλαδή, ε, το λογισμικό ήδη έχει όλες τις πληροφορίες. Μπορείς να έχει πολύ πιο πλούσια δεδομένα ε, ηλεκτρονικά. Γιατί τα τέλη, α, όχι, συγγνώμη, για τους φορτιστές των ε, κινητών τηλεφων, τηλεφώνων, ε, αυτό δεν το καλύπτει η πρόταση τεχνικά. Αλλά νομίζω ότι έφερε αυτή την ε, Επιτροπή, γι' αυτό καλό θα ήταν να το πούμε αυτό με κομψό τρόπο στην Επιτροπή, ούτως ώστε να το α, ε, λάβει υπόψη. Ο κ. Σταγιάννη ασχολείται με αυτό Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μάντρες θα υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε διαφορετικό τρόπο αργότερα. Το τελευταίο σημείο και θέλω να ακούσω και τις απόψεις κομισιών. Υπάρχουν θέματα που αφορούν τους καταναλωτές. Θέματα παρεμβολών. Ε, σε ένα κομμάτι του φάσματος. στα τηλέφωνα τρίτης γενιάς, τετάρτης γενιάς. σας πω ως μηχανικός. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία που καθορίζουν ε, τη συχνότητα στην οποία λειτουργεί το μηχάνημα. Ε, συχνά δεν είναι τόσο υψηλής ποιότητας και δεν είναι... Ε, το διάγραμμα δεν είναι τόσο σαφές, δηλαδή ε, επιτρέπει πολλές παρεμβολές. Υπάρχει η οδηγία EMC, η οποία παίζει ρόλο εδώ και ρυθμίζει τα θέματα καταναλωτών. Ε, δεν χρειάζεται λοιπόν εμείς στην παρούσα πρόταση να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα ε, με τις επιμέρους λεπτομέρειες τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε ε, μεταξύ ημών, οι σκιώδεις συζητητές. Δεν χρειάζεται κατά ανάγκη δηλαδή, να υποβάλουμε και τροπολογίες. Νομίζω ότι όλοι ώστε να μιλήσουν μίλησαν. Η κυρία Λεγκρίπ θέλει να πάρει το λόγο και σε αυτό το σημείο. Όχι. Ο κύριος ε, Τζεράου μπορεί να απαντήσει, να αντιδράσει και αυτός ο πλευράς Κομισιόν στην πρόταση Βάιλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητά και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σχολιάσω την έκθεση Βάιλερ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της, γιατί πραγματικά ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση των στόχων της αναθεώρησης αυτής της νομοθεσίας, δηλαδή θέλει να βελτιώσει τη συμμόρφωση των προϊόντων ε, που καλύπτονται από την οδηγία με, τα, με τις νομοθετικές διατάξεις και τις νομοθετικές απαιτήσεις και σκοπό έχει να απλοποιήσει και το νομικό πλαίσιο. Έχουμε δύο ανησυχίες και κάποιες μικρολεπτομέρειες για ορισμένες τροπολογίες. Αυτά θα επικεντρωθώ σήμερα. Οι ανησυχίες μας αφορούν φυσικά το πεδίο εφαρμογή και το, την καταχώρηση σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Λαμβάνοντα υπόψη και το διδακτικό και το αιτολογικό, έχουμε τι τις τροπολογίε 1, 2, 4, 16, 24, 84 και 87. Κατά τη γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τροπολογίε παρατείνουν το πεδίο εφαρμογή οδηγίες για να, να περιλαμβάνει και του δέκτε και απ' την άλλη το περιορίζει σε συσκευές με δυνατότητες ε, τηλεπικοινωνίας. Που σημαίνει ότι βιομηχανικά και επιστημονικά ιατρικά, ε, επιστημονικές ιατρικές συσκευές αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε την πρόταση, είχε στόχο να τροποποιήσει τον, το πεδίο εφαρμογή και είτε να, να περιλάβει είτε να αφαιρέσει τους δέκτες. Και οι δύο δυνατότητες ήταν ανοιχτέ. Τελικά η επιλογή μας ήταν η πιο απλή, η λιγότερο επαχθής ή αυτή που προβλέπει καλύτερη κατανομή του βάρους μεταξύ των ενδιαφερομένων. Οπότε για τους δέκτες που δεν δημιουργούν εκπομπές, για τους καθαρούς δέκτες, νομίζω ότι ένα μεγάλο τμήμα θα μπορεί να αφαιθεί στα οικειοθελείς, στις οικειοθελείς προδιαγραφές ή στους κατασκευαστές. Οπότε αν πρέπει να λάβουμε υπόψη τους παραμέτρους των, τις παραμέτρους των δεκτών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε στα πλαίσια της οδηγίας EMC. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομικό πλεονέκτημα του προτινόμενου από εμάς πεδίου εφαρμογή είναι ότι με το δικό μας πεδίο εφαρμογή καλύπτουμε όλα τα προϊόντα που δημιουργούν εκπομπές και εσκεμμένα περιορίζουν το ραδιοφάσμα και περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά τα προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τις τον αποκλεισμό των βιομηχανικών, επιστημονικών και ιατρικών συσκευών, προσπαθούμε να προλάβουμε τις ε, μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, γιατί ε, ε, η ασύρματη φόρτιση μας δημιουργεί κάποια προβλήματα, όχι μόνο για τα smartphones και τα κινητά, κυρίως ε, μας ενδιαφέρει η ασύρματη φόρτιση των ηλεκτρικών ε, οχημάτων που μπορεί να είναι πραγματικά μια πολύ ισχυρή φόρτιση, ασύρματη, που μπορεί να ασκήσει παρεμβολές στη χρήση και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε εδώ έναν ε, σαφέστατο κίνδυνο παρεμβολής και να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα. Αν το πεδίο εφαρμογή περιοριστή τη τηλεπικοινωνία, θα πρέπει και αυτές να τις ορίσουμε από νομική άποψη. Γιατί μπορεί να μην είναι σαφέ από νομική άποψη αν μια, η ασύρματη φόρτιση εμπίπτει στον ορισμό της τηλεπικοινωνίας ή όχι. Σε ό,τι αφορά την καταχώρηση το Μητρό, τροπολογίες 6 και 27. Στις προπαρασκευαστικές εργασίες ε, είχαμε διαβουλεύσεις ε, και ακούσαμε τα επιχειρήματα και υπέρ και κατά του Μητρώου. Το Μητρό αποτελεί ε, απέτηση των αρχών εποπτείας αγοράς και χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε ο μηχανισμός αυτός να ενεργοποιηθεί τέσσερα χρόνια μόνο μετά τη θέση σε ισχύ της σχετικής νομοθεσίας. Και λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία των μέτρων που προβλέπονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, αν παρόλα αυτά και μετά την εφαρμογή ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν προϊόντα που δεν ε, συμβιβάζονται με, τα, με τις ουσιώδεις ε, προδιαγραφές, τότε οι αρχές ε, εποπτείας αγοράς θα μπορούσαν να έχουν ένα εργαλείο επιπλέον εξαίρεση που θα είναι αυτό το μητρό. Βέβαια θα έχουμε για κάτι τέτοιο για την εφαρμογή του ευρύτερη διαβουλεύση και με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερόμενους. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι τα παράπονα για το φόρτο, το επιπλέον φόρτο εργασίας που θα επιφέρει στους βιομηχάνους. Όταν έχουμε μαζική μη συμμόρφωση, αυτοί που πλήττονται κυρίω είναι αυτοί που συμμορφώνονται, οι υπάκουοι βιομηχανοί, γιατί το κόστο του Μητρώου είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστο ε, τη συμμόρφωση. Και γνωρίζουμε περιπτώσει όπου οι κατασκευαστέ ουσιαστικά εξοβελίστηκαν από την αγορά εξαιτία του αθέμητου ανταγωνισμού προϊόντων που δεν συμμορφώνονταν με τι προδιαγραφές. Επιπλέον στι Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε συστηματική καταχώρηση των προϊόντων αυτών. Οπότε, αν πάτε στην ε, Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για να ελέγξετε δημόσιες πληροφορίες ε, για την καταχώρηση και το Μητρό, αυτό αρκεί. Και θα έλεγα μάλιστα ότι σε πολλές περιπτώσεις το μόνο βάρος είναι μια επιπλέον ε, διέθεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι μια πλέον διάθεση από αυτή στην οποία στέλνονται ε, οι αιτήσει. Αυτό είναι το μόνο επιπλέον άχθος, η μοναδική επιπλέον υποχρέωση. Θα δούμε στο μέλλον ε, τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στο μέλλον στην ενεργοποίηση της καταχώρησης. Δεν μιλούμε για συστηματική καταχώρηση λοιπόν του εξοπλισμού ή των συσκευών. Μόνο όταν πραγματικά έχουμε ε, κατάφορες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ενεργοποιείται μηχανισμός. Τώρα, κάποιες λεπτομέρειες για τις τροπολογίες. Άρθρο για την ελεύθερη κυκλοφορία, τροπολογία 29. Εκεί προτείνεται απόσυρση του δικτύου ασφαλείας και να εξασφαλίζεται ελεύθερη κυκλοφορία εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οδηγίας. Σε σχέση με τις αντίστοιχες ε, προ... Χρειαζόμαστε αυτή την παραπομπή γιατί ίσως το προϊόν πρέπει να πληρεί και άλλες νομοθετικές διατάξεις όπως περιβαλλοντικές. Οπότε, αν πληρεί τις προϋποθέσεις της, του ραδιοξοπλισμού αλλά όχι τις περιβαλλοντικές, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Χρειάζεται λοιπόν και η παραπομπή. Τόσο ό,τι αφορά τις απαιτήσει υγείας και προστασίας με βάση την οδηγία EMC και για το φάσμα του ραδιοεξοπλισμού που εκπίπτει από την οδηγία EMC. Δεν το συμπεριλάβαμε αυτό γιατί η οδηγία EMC προβλέπει ότι τα προϊόντα που εμπίπτουν στην οδηγία ραδιοεξοπλισμού αποκλείονται. Οπότε στην οδηγία EMC έχουμε αναφορά της οδηγίας χαμηλής τάσης, γιατί η οδηγία LVD χαμηλής τάσης δεν προβλέπει τέτοια εξαίρεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον, την αποκλεισμό υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στο ΙΝΛΕΦ, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε μια οριζόντια συμφωνία που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 32 και 40, εκεί αναφέρεται ότι η απλή δοκιμή για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς καθώς και τους διανομής θα πρέπει να γίνεται μετά με τη ολογημένη αίτηση των αρχών εποπτείας της αγοράς. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο NLF. Για τον το λόγο ότι έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί με τις απλές δηλώσεις συμμόρφωσης και την εποπτεία της αγοράς και οι οικονομικοί τελεστές ε, κανονικά είναι υπεύθυνοι και οι ευθύνε τους ε, ε, εναρμονίζονται με το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι το μόνο μέρος που έχουμε τόσα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά μόνο με απλή δήλωση συμμόρφωσης. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μετάφρασης της ευρωπαϊκής δήλωσης συμμόρφωσης, με βάση την ομοθεσία μας θα πρέπει μια τέτοια δήλωση να συνοδεύει τα προϊόντα. Και το γλωσσικό καθεστώς είναι αυτό που ισχύει συνήθως και που καθορίζεται από τα κράτη-μέλη που έχουν τη δυνατότητα να ζητούν αυτή τη δήλωση στην γλώσσα της, τη δική τους. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 66, ένα άλλο θέμα ουσιαστικά ε, αντιγράφεται πιστά το άρθρο 6. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, γιατί η σχετική διάταξη ήδη καλύπτεται από το άρθρο 6. Υπάρχει και το θέμα του αποκλεισμού του εξοπλισμού ε, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Θα περιμένουμε όμως να δούμε ποια θα είναι η έκβαση των συζητήσεων για το NLF και να το μεταφέρουμε στις οδηγίες EMC και τις σχετικές οδηγίες. Πάντως, αν έχουμε εξαίρεση, θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Γιατί πλήρης εξαίρεση σημαίνει ότι το κάθε κράτος μπορεί, δύναται να έχει δική του νομοθεσία για εξοπλισμό έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, αν ε, τέτοιο εξοπλισμός αποκλείεται πλήρως από τις εναρμονισμένους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας και είναι πρόθυμη να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διευκολυνθεί η λήψη δύο οργανικής συμφωνίας για την νομοθεσία αυτή. Δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση και διαφορά απόψε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε θεωρούμε ότι και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταλήξουμε σε ταχεία συμφωνία για αυτή την νομοθετική πρόταση. Σας ευχαριστώ. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Βάιλερ και πάλι για να σχολιάσει αν θέλει και να συστήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα δεν το έχω, πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Ίσως μπορεί να μας βοηθήσει η γραμματεία. Ε, πάντως, ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή. Μας διατυπώσατε μια-δυο φορές τουλάχιστον την καθεμία της επιφυλάξης σας με κάθε τρόπο και υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να επισημάνω και το έχω προτείνει και με τη συστήση με τους Κιώδης. Ε, έχουμε δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη από ό,τι φαίνεται προς το σύστημα της καταχώρησης σε σχέση με σας. Επομένως, εάν τώρα εσείς μας λέτε ότι Θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική λύση με άλλη μορφή. Φερρυπίν ε, το να ε, δίνεται ένα νέο νούμερο φάξ, τότε σε σχέση με αυτό που προτείνατε αρχικά, το πιο ε, δίσκαμπτο σύστημα, μπορούμε νομίζω να βρούμε λύσεις. Μπορούμε να το συστήσουμε. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να συζητήσουμε όταν υπάρχουν και όλες οι τροπολογίες έτοιμες για να δούμε πώς μπορούμε να τις συνοψίσουμε και πού μπορούμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις που δεν θα είναι βέβαια αντιφατικές μεταξύ τους. Και είναι πολύ σημαντικό με το σύστημα αυτό της καταχώρησης και εάν έχουμε για τα ιατρικά κάποια στοιχεία και μπορούμε να τα δώσουμε, τότε μπορούμε ασφαλώς να προσδιορίσουμε κάποιους κανόνες ώστε να μην κινδυνεύουμε να εισάγουμε μέτρα ή εξελίξεις που θα θέλαμε από την πίσω πόρτα. Παρά τα, όσα είπε, παρά η Επιτροπή, επιμένω ότι δεν χρειάζεται να διεξαχθεί δημόσια κρόαση, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε πώς έχουμε προγραμματίσει τις τροπολογίες μας και κατά τη συνάντηση αυτή, τη συνεδρίαση δηλαδή την επόμενη, πάλι να ξανασυστήσουμε το θέμα με την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν υποθεί και συνδυάζοντας τις λύσεις. Ίσως μπορεί η γραμματεία να μας πει αν έχει τα στοιχεία έτοιμα, τις προθεσμίες, ημερομηνίε κτλ. Ο Πρόεδρος. Εξέταση τροπολογιών, μάλλον προθεσμία 5 Ιουνίου για τις τροπολογίες, για τους σκιώδεις και μέλη της Επιτροπής. 8-9 Ιουλίου εξέταση τροπολογιών πριν το καλοκαίρι, με τις εκοπές Μετά άλλη εξέταση στα τέλη Σεπτεμβρίου και ψηφοφορία τον Οκτώβριο. Επομένως νομίζω ότι έχουμε χρονικό περιθώριο ευρύτατο. Και εσείς αποφασίστε πόση συζήτηση θέλετε να αφήσετε, την περιθώριο συζήτησης με το Συμβούλιο για, το, για την πρόοδο σε επίπεδο Συμβουλίου του θέματος. Ναι και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα αποφασίσετε εσείς, οι σκιώδεις κτλ. Αξίζει τον κόπο νομίζω. Να συνομιλήσετε και με τη Λιθουανική Προεδρία η οποία από ό,τι γνωρίζω έχει αρχίσει να ασχολείται με το θέμα. και ασχολείται ιδιαίτερα και με τα θέματα της ψηφιακής οικονομίας η Λιθουανική Προεδρία. Συμφωνείτε. Καλώς, πολύ ωραία. Έτσι κλείνει το θέμα αυτό. Έχουμε ένα μικρό περιθώριο χρόνου, αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι. Γιατί βλέπω ότι μεταξύ έχει έρθει όλη η ομάδα μας για το θέμα. Κυρία Λεγκρή, εδώ. Να δω, είμαστε όλοι εδώ. Για το 14... Η Επιτροπή είναι εδώ, έτσι. All right, okay. Well, if everybody is happy, I think we can make, uh, we can start early. Uh, which may τα ξεκινάμε λίγο νωρί. Μπορεί να πιούμε και ένα καφέ νωρίτερα, αλλά έχουμε άλλε δεσμεύσει για μετά. Κυρία Βάιλερ, συμφωνείτε με όλα αυτά, δεν έχετε αντίρρηση και προχωρώ. Τώρα, είμαστε στις δύο γνωμοδοτήσεις που έχουμε για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ιατρικός εξοπλισμός in vitro, διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αυτός είναι ο σωστός ο όρος περίπλοκων. Κύριε Σκορέντε Κάμπος είναι Σκιώδη, η κυρία Παρβάνοβα που ήταν εδώ αλλά εξαφανίστηκε, δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσει. Κυρία Ρούλε είναι εδώ, εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Φόξ αν δεν απατώμε. Για να δω. Θα κάνω τι μπορώ με τις προτάσεις του κύριου Φόξ όταν έρθει η ώρα. Εν τω μεταξύ όμως... Ας ακούσουμε την κυρία Λεγκρίπτ και την κυρία Μπέρα, που εκπροσωπεί μάλλον την κυρία Μπέρα, και η κυρία Λεχνιέ και η κυρία Σπανού είναι εδώ. Τις βλέπω πίσω να κάθονται στην τελευταία σειρά. κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συγκεντριά μας, η κυρία Νόρα Μπέρα, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα, γιατί έχει ανοιγμένες υποχρεώσεις ε, πρότερες. Ζητά συγγνώμη από τους συναδέλφους. Η κυρία Μπέρα είχε το χρόνο όμως να διατρέξει τις πολυάριθμες προτάσεις τροπολογίας που έγινε και εξ ονόματός της ε, θα σας, στέλνω το κάτωθι μήνυμα. Η συγκέντριά μας θέλει να ευχαριστήσει πολύ θερμά όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το κείμενο αυτό, με τα κείμενα αυτά. Τους ευχαριστεί για τη θαυμάσια δουλειά της. Οι περισσότερες τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν είναι απόλυτα σκόπιμες και δεν υπάρχουν πολλές δυσκολίε κανονικά για να προσπαθήσουμε να εκπονήσουμε συμβαστικές τροπολογίες, τροπολογίες δηλαδή σύγκλησης. Η κυρία Μπέρα θέλει να κάνει τα εξή σχόλια για κάποιε από τις προτάσεις που κατά την άποψή τη μπορούν να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα ή χρειάζονται κάποιε προσαρμογέ. Για τι ιατρικέ συσκευέ, καταρχά. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή του. Η εισηγήτριά μα εγκατέλειψε την ιδέα του προσδιορισμού των καλοπιστικών αυτών συσκευών, γιατί μπορεί να υπάρχουν παρεμβολές με τα καλλιτικά. Ήθελε όμως να κάνει κάποια διευκρινήση για να καλύψει το α, προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην λιποδιάλυση. Σε ό,τι αφορά τους ορισμούς. Ο κ. Βάμπ έχει καταθέσει μια τροπολογία που προτείνει ένα ορισμό της έννοιας της ασφάλειας. Η τροπολογία 101 που βασίζεται στην απουσία απαράδεκτου κινδύνου. Για την κυρία Μπέρα είναι δύσκολο να εισαγάγουμε έναν ορισμό για ένα τόσο λεπτό θέμα, γιατί μπορεί να ασκηθούν κριτικές για το κατά πόσο κατάλληλο ή κατά πόσο σκόπιμο. Το παράρτημα 1, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ε, λέει πολύ σαφώς πώς εξασφαλίζει η ασφάλεια ενός τέτοιου προϊόντος, μιας συσκευής. Η συγκήτριά μας δεν πιστεύει ότι μπορούμε να μιλήσουμε για αποτελεσματικότητα εντό αγωγικών για ένα προϊόν, όπως προτείνεται στην τροπολογία 102 από την κυρία Παρβάνοβα. Αν αυτή η έννοια δεν έχει ήδη οριστεί πιο πάνω. Όμως ένας τέτοιο ορισμό είναι σύνθετος, δύσκολο να γίνει. Πώς θα ορίσουμε ας πούμε, την αποτελεσματικότητα μιας, αναπνευστικής, μιας αναπηρικής καρέκλας ή ενός απεινιδωτή θα προτιμούσε να μιλήσει για, κλινική, για κλινικά ωφέλη, αν σας διευκολύνει αυτή η έννοια. Η κυρία Μπέρα επίσης υποστηρίζει την έννοια της επίδοσης που προτείνει ο κ. Κορέι, Αντεκάμπος στην τροπολογία 105. Η έννοια της επίδοσης είναι ουσιαστική για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υπάρχει σε όλο το κείμενο, γι' αυτό που καλό είναι να ξεκαθαριστεί τι σημαίνει σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των operators. Η κυρία Μπέρα αναφέρει στις τροπολογίες της κυρίας Βάις Κέρμπερ 115 και 118. Θεωρεί ότι πρέπει να κολλήσουμε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τις ε, ευθύνε των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των διανομέων. Για λόγους ασφάλειας, η συγκήτρια δεν θέλει να αμφισβητήσει τις αρμοδιότητες και ευθύνε του καθενός. Καταλαβαίνει τις δυσκολίες που υπάρχουν προς τη διαχείρισή τους, που μπορεί να, δημιουργεί, να δημιουργήσουν αυτές οι διατάξεις σε κάποιου φαρμακοποιού, αλλά θα προτιμούσε η Κομισιόν να κάνει τι προσαρμογέ ανά περίπτωση για ορισμένα επαγγέλματα, αν χρειάζεται. Τώρα, για την υποχρέωση ε, που προβλέπει το άρθρο 116 τη πρόταση του κανονισμού. Η κυρία Μπέρα συμφωνεί να αποκλείσουμε κάποια προϊόντα όπως οι αγράφες ή ε, τα οδοντιατρικά σφραγίσματα. Θα, ήθελα, θα ήθελε να μας πει η Κομισιόν την άποψή της ε, για τις, τα ορθοπαιδικά, τις ορθοπαιδικές προσθήκες. Στι 124, ε, τροπολογία 124 ζητάμε από την Κομισιό να δει ένα περίπτωση τι μπορεί να εξαιρεθεί από αυτήν την υποχρέωση. Σε ό,τι αφορά την, το περιεχόμενο αυτών των χαρτών θα πρέπει να μην βάλουμε τις μη απαραίτητε πληροφορίε ή πληροφορίε που δεν χρησιμοποιεί ο ασθενής, ώστε να μην ε, βάλουμε πολύ άχθος ό,τι αφορά την δήλωση ε, συμμόρφωση ε, τροπολογίες 128 και 129. Η συγκήτριά μας θέλει να παραμείνουμε στις υποχρεώσεις ε, του νέου νομοθετικού πλαισίου που είναι σαφής και που, με βάση το οποίο κάθε πολίτης και κάθε επαγγελματία της υγείας μπορεί να γνωρίζει στη γλώσσα του ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Σε ό,τι αφορά τους ε, κοινοποιημένους οργανισμούς, η πρόταση του συναδέλφου μας, του κυρίου Φόξ, η συγγήτριά μας ε, υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν που θέλει να πλαισιώσει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων αυτών οργανισμών. Πιστεύει ότι είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να μπορούν να αμφισβητούν μια κοινοποίηση αν το θεωρούν σκόπιμο. Και η Κομισιόν θα πρέπει να δίνει την άποψή της και να, στα... να προκαλέσει αναστολή αυτής της κοινοποίηση. Παραδείγματο χάρη, σε τεχνητά μέλη, ε, χάρη του ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, για τις συσκευές κινδύνου. Δεν υπήρξαν εναλλακτικέ προτάσεις για αυτό το σημείο. Ο κύριος Βάμπ προτείνει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες στις, στους ελέγχους των κοινοποιημένων οργανισμών. Αυτή η προσέγγιση όμως, κατά την εισηγήτριά μας, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, που είναι και η Κομισιόν νομίζω συμφωνεί, να πλαισιώσουμε διαφορετικά την θέση στην αγορά των ε, καινοτόμων ε, προϊόντων. Η συγγήτριά μας θέλει να υπενθυμίσει ότι άκουσε όλους τους, ενδιαφερο... όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο, ώστε να κάνει μια επικοδομητική πρόταση που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ε, κατασκευαστών και των ενώσεων των ασθενών και καταναλωτών. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα μακροπρόθεσμα, εναρμονίζοντας τις πρακτικές, χωρίς όμως να προσθέσουμε περιτές προθεσμίες που δημιουργούν προβλήματα ε, στους κατασκευαστές, γιατί το φοβούνται πραγματικά αυτό οι κατασκευαστές. Επίσης, οι συστάσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές ε, για το αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήρια για την αξιολόγηση από τους Ευρωπαίους ε, εμπειρογνώμονες. Και αν αυτό θα δώσει δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές, στους κοινωνικοποιημένους οργανισμούς και στα κράτη-μέλη να φτιάξουν αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, ούτως ώστε να έχουμε συγκλίνουσες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα πραγματικά καινοτόμα προϊόντα θεωρείται η εισηγήτριά μας ότι χρειάζεται να δοθεί μια ανεξάρτητη γνώμη. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για τα για τους ματοδότες, για τα στέντ και τα που εύκολα πλαισιώνονται από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά μιλάμε και για τις ε, καρδιακές βαλβίδες ε, που μπαίνουν υποδόρια, για στέντ ε, που περιβάλλονται από μια φαρμακευτική ουσία, για ανιχνευτές που μπαίνουν στην καρδιά και Μιλάμε για καινοτόμε δηλαδή συσκευέ. Όποια και να είναι η γνώση των εμπειρογνωμών και των κοινοποιημένων οργανισμών, η θέση στην αγορά αυτών των προϊόντων θα πρέπει να αξιολογεί από μια ανεξάρτητη αρχή που έχει πραγματικά στο εσωτερικό τη την απαραίτητη ε, πραγματογνωμοσύνη. Χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών για τόσο καινοτόμα προϊόντα. Δεν χρειάζεται μια και μόνο ε, πραγματογνωμοσύνη, αλλά περισσότερε ε, στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την διαφάνεια για τις κλινικές έρευνες, ο κύριος Κορέι Κάμπος έχει καταθέσει πολλές ε, τροπολογίες για την ε, δημόσια πρόσβαση. Άρθρο 151, σε πληροφορίες εννοώ. Ε, φυσικά η κυρία Μπέρα θέλει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, αλλά θέλει να μην δημοσιεύονται αφιλτράριστα τα στοιχεία, τα δεδομένα. Πρέπει να είμαστε συνετοί σε αυτό το σημείο και θεωρεί ότι η πρόταση της Κομισιόν πηγαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Ε, έχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε αναπερίπτωση τις πληροφορίες που μπορούν να δημοσιοποιηθούν ή όχι. Δεν είναι οι κατασκευαστές, αλλά η οχι δεν ειναι οι κατασκευαστε αυτή που αποφασίζει πότε δίδεται πρόσβαση σε αυτέ τι πληροφορίε και πότε όχι. Επίση, κατά τα λοιπά, για τι έρευνε. Ε, τα σχετικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να αποστέλλονται στην, στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβούλευση με την Επιτροπή Διοντολογίας. Δεν θέλω να... Η συγκεκριά μας δεν θέλει να απομακρυνθούμε πολύ από αυτό που υιοθε... υιοθετήθηκε από την... τον πρόσφατο κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές. Για τους κανόνες ε, ταξινόμησης. Ο κ. Σβάμπ έκανε προτάσεις για να αποκλείσουν ορισμένα προϊόντα κυρίως χειρουργικό υλικό από την κατηγορία 3. Η συγκίτριά μα ε, για λόγου αρχή δεν αντιτίθεται, αλλά θέλει την άποψη τη Κομισιόν για το σημείο αυτό, για να εξασφαλίσει ότι δεν αποχαρακτηρίζουμε προϊόντα τα οποία ενέχουν πολλού κινδύνου παρόλα αυτά. Πολλέ τροπολογίε είχαμε για τι καταξιδότητε πράξη. Η συγκίτριά μα λέει πρέπει να το δούμε αυτόν ο περίπτωση. Ορισμένοι θέλουν να περιορίσουν και να προσφεύγουμε στην τακτική νομοθετική διαδικασία όσο να τον περισσότερο. Η συγγήτριά μα λέει ότι πρέπει να κρατήσουμε του κανόνε επιτροπολογία και να κάνουμε προσαρμογή αν χρειάζεται. Δεν έχει προβλήματα επί τη αρχή ε, αυτού, αλλά θέλει να ακούσει την άποψη των αρμοδίων νομικών υπηρεσιών πριν αποφασίσει. Κατά τα λοιπά, όπω είπα και στην αρχή, η συγγήτριά μας θεωρεί ότι πολλέ από τις ε, προτάσεις και συστάσεις των συναδέλφων είναι πολύ σκόπιμες. Οι προτάσει του Κορέντε κάπω και παρά, ε, της κυρία Παρβάνου για την ε, επαναχρησιμοποίηση είναι πολύ σωστέ. Για τα οριακά προϊόντα, οι προτάσεις κυρίας Παρβάνοβα 108 και 109, το να προσφύγουμε σε εμπειρογνώμονες που έχουν ποικίλε γνώσεις, είναι πολύ σωστή. Πρέπει να μα δώσει η Επιτροπή τη γνώμη της για το κατά πόσον γίνεται κάτι τέτοιο. Τελευταίο κεφάλαιο. Το in vitro διαγνωστικό Τεχνολογικό προϊόν. Σε ό,τι αφορά την ε, α, παρέκκληση της κατηγορίας D. Ε, θα πρέπει να βρεθεί συμβιβασμό, λέει η συγκεκριμένη με τον κύριο Φόξ. Η κυρία Μπέρα θέλει να υπενθυμίσει ότι έχουμε διαφορετικές επιδόσεις στην Ευρώπη για κάποια προϊόντα τάξης ε, κατηγορίας D in-house. Εν συνεχεία πρέπει να βάλουμε όρια. Δεν θα πρέπει οι μαθητευόμενοι μάγοι δηλαδή να μπορούν να φτιάχνουν τα δικά τους ε, μηχανήματα χωρίς κανέναν έλεγχο. Θέλει λοιπόν να Διευρυθεί αυτή η παρέκκληση σε κάποια μηχανήματα της κατηγορίας D, αλλά θέλει να βρεθεί μια ισορροπία όμως, ούτως ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή εγγύηση ασφάλειας. Καταληκτικά. Η συγκήτριά μας ευχαριστεί ακόμα όλους όσους και όσες τροφόδωσαν τη συζήτηση και έκαναν προτάσεις. Πιστεύει ότι μπορούμε να βρούμε συμφωνία σε όλα αυτά τα σημεία και θα προτείνει όσον ούπο μία συνεδρίαση με τους κοιόδους και φυσικά το γραφείο της κυρίας Μπέρα είναι στη διάθεση και των σκιωδών εισηγητών και των υπολείπων ευρωβουλευτών που έχουν ερωτήσεις που θέλουν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που αντικαταστήσετε την εισηγήτρια με πραγματικά απάξιο τρόπο. Ας ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις ηγητές. Ο καθηγητής Κορέα Δεκάμπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ φυσικά να συγχαρώ την συνάδελφο Νόρα Μπέρα για την τεράστια προσπάθεια που έκανε αναλύοντας αυτές τις δύο προτάσεις και συντάσσοντας ε, τις δύο γνωμοδοτήσεις της. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το έργο της εισηγήτριας και προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να τελειοποιήσει αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις. Πιστεύω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια ενιαία και καλή πρόταση. Οι τροπολογίες, ε, ας μην ξεχνούμε, ότι θέλουν να ενισχύσουν, κυρίως στην δική μας Επιτροπή, να ενισχύσουν την διαδικασία πιστοποίησης και παρακολούθησης των ε, διαφόρων ε, συσκευών ιατρικών στην ευρωπαϊκή αγορά για να ενισχυθεί η ασφάλεια για τους καταναλωτές. Και φυσικά αυτό θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Συμφωνούμε με όλες τις προτάσεις που θέλουν να ενισχύσουν ε, τις αρμοδιότητες των επιστοποιημένων οργανισμών, των κοινοποιημένων οργανισμών και μάλιστα μόνο ορισμένες, ορισμένοι θεροκισμένοι κοινοποιημένοι οργανισμοί που υπακούν σε κάποια κριτήρια μπορούν να οδηγήσουν στην έγκριση ε, ιατρικών συσκευών ε, μεγάλου, υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν αρμοδιότητες ε, στον κλινικό τομέα για έναν πιο εδελεχή και αυστηρό έλεγχο των κλινικών δοκιμών και αξιολογήσεων που γίνονται από τους Κατασκευαστέ, που είναι και το αδύναμο σημείο του, και το πιο τροτό σημείο του συστήματος. Επίση θα πρέπει να ενισχύσουμε τους κοινοποιημένου οργανισμούς απέναντι στους κατασκευαστέ, τους παρασκευαστές επιβάλλοντα υπεχωρατικούς, ε, τυχαίους, ε, δημοτοληπτικού ελέγχους. Χαίρομαι για τις τροπολογίες που ζητούν καλύτερο έλεγχο ε, των κοινοποιημένων οργανισμών και τονίζουν την ανάγκη ισχυρότερου συντονισμού και μεγαλύτερης συνεργασίας των αρμόδιων εθνικών αρχών με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την πραγματοποίηση κοινών ελέγχων και επιθεωρήσεων από μία και παραπάνω αρμόδιες αρχές για καλύτερη πρόσβαση στις στην ενιαία αγορά και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. Σε δύο τομείς ε, που σημαντικούς θέλουμε ενίσχυση της ε, διαφάνειας και της ποιότητας των κλινικών δοκιμών και των, της παρακολούθησης ε, του ιστορικού χρησιμοποίησης των ιατρικών συσκευών μετά την εισαγωγή του στην εσωτερική αγορά. Γιατί είναι πολύ διαφορετική αυτή η αγορά από την αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων. Γι' αυτό και το Μητρό Ιστορικού αντικαθιστά κάτι που ήταν αδύνατο με τα φάρμακα. Γιατί μερικές φορές έχουμε διπλές τυφλές κλινικές δοκιμές. Χρειάζονται τέτοιου είδους δοκιμές για τέτοιο εξοπλισμό, ιατροτεχνολογικό και τέτοια προϊόντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ενιαίο μηχανισμό πιστοποίησης, ταυτοποίησης και κεντροποιημένη βάση δεδομένων, είναι βασικό στοιχείο της νέας διαδικασίας, γιατί το μητρό του ιστορικού είναι πολύ σημαντικό, αλλά και το τελευταίο σημείο είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος. Σε ό,τι αφορά τους, κλινικέ τις κλινικές δοκιμές που προηγούνται ή συνοδεύουν την θέση εμπορία, μέχρι στιγμής ήταν πολύ αόριστες αυτές οι δοκιμές και μη δεσμευτικέ. Θέλουμε ενίσχυση αυτών των ελέγχων για αύξηση της ποιότητας και της διαφάνειας. Επίσης, πρέπει να γίνονται έλεγχοι και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κάτι που είναι απαραίτητο για σωστό έλεγχο των δεδομένων αυτών, για να μπορέσουμε να δείξουμε νέες διαδικασίες ε, αυτοματοποιημένης ε, επιτήρησης, με βάση την κλινική εμπειρία που έχουμε. Η, η συμφωνεί με τον έλεγχο αυτό, που είναι εντελεχέστερος, θεωρεί όμως ότι πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο για τον έλεγχο αυτό και αυτό το φίλτρο ε, να είναι ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι και απαιτητικοί στο τομέα αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία στο τέλος. Επίσης αυτός ο μηχανισμός σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια υγεία θα προβλέπει έγκαιρη προειδοποίηση κάποιων ε, ανησυχητικών ε, δειγμάτων, ιδιαίτερα όταν έχουμε μεγάλο αριθμό ασθενών που επηρεάζεται και επίσης είναι σημαντικό να είναι προσιτό το ιστορικό ώστε όλοι έχουν, όλοι έχουν πρόβλημα να μπορούν να στέλνουν την κοινοποίησή τους, ε, την επισήμανση και να μπορούμε να έχουμε ε, σε πρόωρο στάδιο ανάκληση του προϊόντος αυτού. Επίσης θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη χρήση νέων ε, συσκευών σε σχέση με τις παλιές ώστε να ενισχυθούν και τα εθνικά συστήματα και η αποδοτικότητα των εθνικών συστημάτων υγείας. Ελπίζω να συμφωνήσει η Γετρία με τις προτάσεις αυτές. Είμαι στη διάθεσή της για περαιτέρω ε, συζήτηση και επεξεργασία προκειμένου να λάβουμε υπόψη το συμφέρον και των ασθενών και φυσικά και της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και αφού δεν υπάρχει κανείς από τους φιλελευθέρους... Α, όχι, έχει έρθει ο κύριος Φόξ. και κυρία Ρούλε, αλλά ο κύριο Φόξ με πολύ στενά. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και στο συγγνώμη που έφτασα κάπως καθυστερημένος. Ξέρετε, ότι είμαστε σε πολλέ επιτροπέ έχουμε τέτοιε δυσκολίε. Ναι, λέει ο πρόεδρο, αλλά αρχίσαμε και λίγο πιο γρήγορα σήμερα, οπότε έχετε τη δικαιολογία σα. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τον συγητή και του Σκιώδης για τη συνεργασία. Θα ήθελα να αναφερθώ στα κύρια θέματα των τροπολογιών. Υποστηρίζω αυτές οι οποίες αλλάζουν τις στην πράξη και τις μετατρέπουν σε κοινή νομοθετική διαδικασία. Μόνο με εφαρμοστικέ πράξει θέλω να γίνεται η εξοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με τι από τι τροπολογίε τι οποίε έχει καταθέσει ο κύριο Σουάβ και Είμαι υπέρ τη θέσπιση μια κεντρική υπηρεσία. Χαίρομαι που ο κύριο Φαπ προχωρεί περαιτέρω των δικών μου προθέσεων για να επικεντρώσει την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ρόλο της ε, ιατρικής υπηρεσίας για την ε, επαλήθευση και τον έλεγχο με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Στις δικές μου τροπολογίες δείχνω ότι ε, διαφωνώ στο να είναι για την ε, κοινή εκθέση αξιολόγηση δεσμευτικές οι θέσεις υπηρεσίας αυτής. Νομίζω ότι μπορεί απλώς να δώσει μια ε, όθηση, ένα κίνητρο για περισσότερο έλεγχο στις αρμόδιες αρχές και όχι να παραδώσει αρμοδιότητες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συμφωνώ λοιπόν με την προσέγγιση αυτή και καλώ τους συναδέλφους ευρωβουλευτές να επιλέξουν αυτήν και όχι την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, η προσέγγιση τη Επιτροπής οδηγεί και σε καθυστερήσει και σε επιπλέον κόστο, χωρί να μας αποδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε ε, περισσότερη ασφάλεια ή εγγύηση για τον καταναλωτή. Σε κάποια σημεία που έχω ανησυχίες, συγκεκριμένα τροπολογία 102, η οποία προσπαθεί να ρυθμίσει την αποκαταλεσματικότητα των ε, μηχανημάτων αυτών, τον, του εξοπλισμού αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που όμως μπορεί μόνο σε επίπεδο πιο κοντά στον ε, ασθενή και δει σε εθνικό επίπεδο, εκεί όπου έχει και το κράτος τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ε, επαλήθευσης για να το βεβαιώσει. Οι τροπολογίες 145-155 μιλούν για κοινοποιημένους οργανισμούς, για γνωστοποιημένου οργανισμούς, με αποτελέσματα όμως πολύ διαφορετικά και δεν βλέπω κανένα λόγο να ε, υπάρξει τέτοιου είδους ε, υπαγωγή και νομίζω ότι πρέπει οι αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την λειτουργία των γνωστοποιημένων οργανισμών μέσα από τις διαδικασίες επαλήθευσης. Καλύτερη διαφάνεια ε, θα σήμαινε βέβαια και καλύτερη προϋποθέτει και καλύτερη εποπτεία στην υπόθεση αυτή. Όσον αφορά τώρα τα in vitro διαγνωστικά τεχνολογικά προϊόντα, συμφωνώ ε, να υπάρχουν έλεγχοι για τις κατηγορίες α έως 10 όταν δεν υπάρχουν, για ε, παραδείγματι για σπάνιες αρρεώστιες ασθένειες και με σημαντική επίπτωση ως προς την διάγνωση που μπορεί να σώσει ζωές. Θα πρέπει να θεσπιστούν λοιπόν από τα εθνικά όργανα οι κατάλληλε διαδικασίε για την ποιότητα και την επαλήθευση των ε, ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η υπηρεσία αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση και ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. Η κυρία Πιέτη Κάινεν θέλει και εκείνη να λάβει το λόγο. Έχει μια σειρά από τροπολογίες. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχάς, έχω μια προσέγγιση γενικά συγγενή με αυτήν του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών ε, περισσότερο. Αυτό που θα ήθελα εγώ να επισημάνω όμως είναι σε ένα θέμα που ίσως να χαρακτηριστεί ελάσσον σε σχέση με το γενικό πεδίο εφαρμογής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αλλά από την ανθρώπινη σκοπιά ίσως να έχει τεράστια σημασία. Και αναφέρομαι στα τεχνητά μέλη. όπως εμφυτεύματα μυρού και εδώ η τυποποίηση τέτοιου είδου τεχνητών μελών μπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, από τον ένα γιατρό στον άλλον, ανάλογα με τον κατασκευαστή του ε, τεχνητού μέλους. Και ενδέχεται να υπάρχει εγκατεστημένο τεχνητό μέλος, αλλά σε κάποιο τμήμα του όταν χρειαστεί κάποια αλλαγή να μην υπάρχει συμβατό ε, τμήμα ε, λόγω διαφορών κατασκευαστικών και προδιαγραφών. Πράγμα το οποίο προφανώς δημιουργεί προβλήματα, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τραυματισμούς, η εισαγωγή του τεχνητού μέλους και καθυστέρηση στην ανάρρωση. Και σας λέω ότι όπως και στο θέμα των φορτιστών για συσκευές φορητές, με τον ίδιο τρόπο, αλλά πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις, εξετάζω και εγώ το θέμα των τεχνητών μελών και βλέπω ότι και η βιομηχανία δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει εσωτερικά. Κάποιες τροπολογίες λοιπόν που καταθέτω ακριβώς αποσκοπούν σε αυτό. για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να συζητήσουμε την τυποποίηση, όποιος είναι ο τύπος, όποιο είναι το πρότυπο στο οποίο θα καταλήξουμε, θα πρέπει η τυποποίηση να αποτελέσει τη βάση για το μέλλον. Και στο την κατανόησή σας και την υποστήριξη σας και αυτή την πτυχή ιδιαίτερα για τα τεχνητά μέλη. Ο Πρόεδρος. Όπως είπα από πλευρά βιομηχανικών και βιομηχανολογικών προϊόντων ίσως υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά αυτά τα τεχνικά μέλη που αναφέρεται, αλλά θα το συζητήσουμε. Γιατί η τεχνολογία προχωρά με ε, τεράστια άλματα σε ό,τι αφορά τα υλικά που χρησιμοποιεί για τέτοια τεχνητά μέλη και φυτεύματα. Και είχα, υπάρχουν άνθρωποι που είχαν φυτεύματα ισχύου ε, για πάρα πολύ καιρό και τώρα χρειάζεται ακόμη και για να να αλλάξουν ε, το, το εφήτευμα αυτό, γιατί στο παρελθόν ε, δεν ε, ζούσαν τόσο πολλοί άνθρωποι, περισσότερο από το, τη διάρκεια ζωής του εφητεύματος, τώρα ζουν πολύ περισσότερο και τα υλικά αλλάζουν. Κύριε Σπανού, θέλετε το λόγο, παρακαλώ, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο και ευχαριστώ και τους Ευρωβουλευτές Πολλά μαθαίνουμε σήμερα. Το πρωί ήμασταν στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος, ε, τώρα το απόγευμα σε εσά και θα πάμε αργότερα στην Επιτροπή Απασχόλησης και μας ε, εντυπωσιάζει ο πλούτος αλλά και η διάσταση απόψεων μεταξύ των διαφόρων τροπολογιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έγκρισης και διοδότησης. Πάντως όλοι θα μάθουμε, θα μάθουμε αυτή τη διαδικασία και θέλουμε όλοι να ενισχύσουμε τη διαδικασία έγκρισης, γιατί στόχος μας είναι η ασφάλεια, το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους Ευρωπαίους ασθενείς. Οπότε, όπως είπαμε και το πρωί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα ήθελα και πάλι να διατρανώσουμε την επιθυμία μας να ενισχύσουμε τα επίπεδα ασφάλειας χωρίς να επηρεάσουμε την ισορροπία της πρότασης. Γιατί η πρότασή μας ε, στόχο δεν είχε την ε, έγκριση πριν τη θέση αγορά. Αυτό φάνηκε και από τη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έδειξε ότι δεν έχει προστιθέμενη αξία με τέτοια πρόορη έγκριση. Αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε τα κριτήρια για του κοινοποιημένου οργανισμού ή την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών. Αυτό περισσότερο μα ενδιαφέρει και αυτέ τι κατευθύνσει ε, θα παροτρύνουμε, θα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι έτσι θα εξυπηρετηθεί η την παρακολουθηση των κοινοποιημενων οργανισμων αυτο περισσοτερο μα ενδιαφερει και αυτε τι κατευθυνσει θα παροτρυνουμε θα ενθαρρυνουμε τα κρατη μελη Πιστεύω οτι ετσι θα εξυπηρετηθει η προταση και θα διδαχθούμε και από τα μαθήματα που αντιλήσαμε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ιατρικών συσκευών. Έχουμε πολλές τροπολογίες που προβλήθησαν από την εισηγήτρια και από άλλα μέλη της Επιτροπής. Μερικές είναι πολύ θετικές και είναι και στη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις κλινικές δοκιμές, για παράδειγμα, που θα, ε, θα πρέπει να είναι πιο πλούσιες. Έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο αυτό για τις κλινικές αξιολογήσεις και έρευνες Φυσικά έχουμε αντίστοιχη πρόταση για τι κλινικέ δοκιμέ, οπότε και οι κλινικέ αξιολογήσει θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτό και να μην ξεχνάμε και τον κανόνα τη εμπιστευτικότητα. Επίσης θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ε, τις, ε, τους τρόπους για τον ιατρο, ιατρο, ιατρολογικό εξοπλισμό και υπάρχουν και διαγνωστικό ιατρο, ιατροτεχνικό εξοπλισμό και επίση, κάτι που προέκυψε από το ρόλο των εμπειρογνωμόνων από πολλούς τομεί, Μερικές τροπολογίες ήταν κάτι τέτοιο, αλλά ίσως είναι ανέφικτη αυτή η πρόταση. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Και αν δεν κάνω λάθος, μιλούμε και για τη δεύτερη πρόταση, τα εξαρτήματα in vitro για το διαγνωστικό ιατροτεχνικό προϊόν. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία Δέλτα που ανέφερε κάποιος ευρωβουλευτής, Όντως, ε, έχει νόημα η εξαίρεση αυτή και σίγουρα η πρόταση χρήζει περαιτέρω εξέτασης. Ελπίζω να καταλάβατε πάνω κάτω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί προωθήσατε με ταχύς ρυθμούς αυτό το θέμα που είναι για μας προτεραιότητα και πραγματικά ευελπιστούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα σε πρώτη ανάγνωση ε, κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Μιλήσαμε για την σημασία της ασφάλειας και προστασίας των ασθενών, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας που έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι προς όφελος όλων να κινηθούμε με ταχύς ρυθμούς και ελπίζω με επικοδομητικό τρόπο και πριν την ψηφοφορία να ολοκληρωθεί η εξέταση και η συμφωνία προς τροπολογίες. Ευχαριστώ. η κυρία Λεγκρίπ φαίνεται ότι αποφάσισε να φύγει. Ας ολοκληρώσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή και όλους όσοι έχουν συμπράξει στο έργο αυτό. Για να δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα για να προχωρήσει ο φάκελος και το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος φυσικά ταυτόχρονα. Συμβαστικές τροπολογίες θα εξεταστούν στις 17 Ιουνίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 18 Ιουνίου η Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 10 Ιουλίου, αν δεν απατώμε. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Οι σκιώδεις ηγητές θα τα κοιτάξουν μαζί με την κυρία Βερά. Και έτσι, ολοκληρώνουμε για σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είχαμε προβλέψει μια συζήτηση για την έκθεση για τις υπηρεσίες, αλλά η κυρία Κοράτσα δεν ήταν ε, διαθέσιμη. Και έτσι σταματούμε τη συνεδρίασή μας μέχρι τι 5 και 4, γιατί μετά θα συνεχίσουμε μόνο με συντονιστέ. Έτσι τελειώνει το δημόσιο τμήμα τη συνεδρίασεώ μα και θα συνεχίσουμε μετά και κλεισμένο των θυρών μόνο με συντονιστέ. Υπενθυμίζω στους συναδέλφου ότι αύριο το πρωί συνεδριάζουμε για ανταλλαγή απόψεων από 9 μέχρι 10 για το ψηφιακό θεματολόγιο με την κυρία Νέλη Κρούς. Μετά τις 10 έχουμε ψηφοφορίες για πολύ σημαντικά θέματα. Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, οδηγία για τον καπνό, παραπλανητικές πρακτικές, οχήματα με κινητήρα και περιμένω να σας δω όλους για την ψηφοφορία στις 10. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους και το κοινό από το διαδίκτυο που μας παρακολουθεί ότι υπάρχει το δελτίο της Επιτροπής μας στη διάθεσή σας. Το έχετε λάβει βεβαίως όλοι στο γραμματοκιβώτιό σας όλοι οι συνάδελφοι, αλλά αν τυχόν το χρειάζεστε υπάρχει στον ιστότοπο της Επιτροπής, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και μπορείτε να το ε, βρείτε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Πέραστε συνεδριά σας και συντονιστές στις 5 και 4.